Καλημέρα σας. Πολύ καλημέρα σας, αγαπητοί συνάδελφοι. Σας καλωσορίζω θερμότατα, όλους εσάς τους πολυαρίθμους παρόντες. Ιδιαίτερα θέλω να καλωσορίσω τους παρόντες, ακριβώς. Γιατί οι άλλοι που θα αργήσουν χάσανε οι καθυστερημένοι. Πάντως θα φροντίσω να αρχίζουμε πάντα στην ώρα μας συνεδριάσεις, έτσι ώστε να έχουμε και τον απαραίτητο χρόνο στη συνέχεια. Έρχομαι τώρα στην ημερήσια διάταξη και σας ερωτώ. Μάλλον να σας προτείνω μία αλλαγή εγώ. Ε, το σημείο 10 θα πρέπει να το αναβάλουμε, γιατί με παρακάλεσε η συνάδελφος Βαλεάν να αναβάλουμε αυτό το θέμα και θα το δούμε στις 5 Οκτωβρίου στις 5.30 ε, το απόγευμα, συμφωνείτε. Gibt es sonst noch Tagesordnung? Α, έχουμε τίποτα άλλο για την ημερήσια διάταξη. Ο Τσάρλς Τσίτσεστερ. Πρόεδρε, λυπάμαι που πρέπει να σας πω ότι τα γερμανικά μου δεν φτάνουν στο να σας ε, καταλαβαίνω πολύ τόσο απευθείας. Αλλά Είχα πρόβλημα με τη διερμηνία διότι άρχισα να ακούω αγγλικά, μετά άλλαξε η γλώσσα, μετά έγινε γερμανικά. Εγώ νομίζω ότι είμαι στο κανάλι. Δεν ξέρω τι έχει μπλέξει εκεί τεχνικά, και ζητώ συγγνώμη, δεν άκουσα το τελευταίο αυτό που είπατε. Ευχαριστώ πολύ. Είναι εντάξει τώρα τα τεχνικά της Ερμηνείας. Ε, Ωραία, να επαναλάβω τότε. Έλεγα ότι το σημείο 10 τη σημερινής διάταξη, επενδυτικά σχέδια σε ενεργειακή υποδομή εντό τη Ευρωπαϊκή Κοινότητα, θα πρέπει να αναβληθεί, διότι με παρακάλεσε η συνάδελφο ε, κυρία Βαλεάν να το συζητήσουμε στις 5 Οκτωβρίου. Εντάξει. 6 Οκτωβρίου. Στις 6 Οκτωβρίου. Α, το άλλαξε πάλι η γραμματεία χωρίς να μου το πει. Οπότε πάει στις 6 Οκτωβρίου. Μπας περιπτώσει για την άλλη εβδομάδα να βάλετε. Συμφωνείτε. Συμφωνείτε. Σημείο 2. Ανακοινώσεις του Προέδρου. Θα ε, ήθελα να επικεντρωθώ στα πρακτικά των συντονιστών της Δευτέρας Σεπτεμβρίου. Ελπίζω να τα έχετε λάβει όλοι και να τα έχετε κοιτάξει κιόλας. Έχει θέματα που έχουν να κάνουν με τις αντιπροσωπείες, ταξίδια, ανάθεση εκθέσεων και παρακαλώ πολιτικές ομάδες να εκδηλωθούν και να ενημερώσουν. Λοιπόν, αν δεν έχετε τίποτα άλλο για τις ανακοινώσεις, πάει και αυτό και πάμε στο σημείο 3. Ευρωπαϊκό πρόγραμμα τηλεπισκόπησης, γεωσκόπησης. Είναι μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αποφασίσαμε εμείς συνειδητά να αφιερωθούμε σε αυτό το θέμα και από σήμερα το συζητήσουμε και χαίρομαι γι' αυτό. Ο συνάδελφος Γκλάντε είναι συγητή. Υποθέτω ότι μιλήσει, θέλει να μιλήσει πρώτος ή πρώτα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Καλά, η Κομισιόν. Γιατί όλα αυτά είναι νέα έγγραφα που μας προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και καλό θα ήταν να μας ενημερώσει για την κατάσταση των πραγμάτων και μετά θα ακούσουμε τον κύριο Γκλάντε και τους κύριους συγητής. Ποιος είναι εδώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αρμόδιος και παρόν. Δεν βλέπω το ονοματάκι σας, λυπάμαι πάρα πολύ. Είμαι ο Είμαι Πολ Βάισενμπεργκ, είμαι ο υπεύθυνο ε, διευθυντή ε, για την ε, δορυφορική πολιτική. Ευχαριστώ πολύ κύριε που μου δώσετε τη δυνατότητα να κάνω μια σύντομη εισαγωγή στην πρόταση που έχετε μπροστά σα. Είναι η πρώτη φορά που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συζητάει την λειτουργική φάση του GMS, του Ευρωπαϊκού Προγράμματο Γεωσκόπηση. Περί τίνο πρόκειται, πρόκειται για ένα σύστημα το οποίο παρέχει πληροφορίες. Και αυτές οι πληροφορίες βασίζονται σε δεδομένα τα οποία παράγονται από μια υποδομή παρατήρησης ε, στο έδαφος, ε, στον αέρα, στην ε, θάλασσα ή στο διάστημα. Αυτό, αυτή η σφαιρική, το σφαιρικό πρόγραμμα παρατήρησης είναι, συνιστά ένα πρόγραμμα γεωσκόπησης το οποίο έχει εκπονήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και το οποίο ε, αφορά ερευνητικές ε, δραστηριότητες τις οποίες συμμετέχουν από κοινού οι χώρες μέλη και η GMS. E Πρόκειται για ένα εργαλείο λοιπόν το οποίο παρέχει συγκεκριμένες υπηρεσίες και θα ήθελα να σας δώσω ορισμένα παραδείγματα. Το GMS e ε, δίδει, παρέχει προστασία στους πολίτες σε περίπτωση πυρκαγιών, πλημμυρών, σεισμών, ένα σύστημα παρατήρησης των ωκεανών και της ε, ποιότητας της ε, ατμόσφαιρας κλπ. Λοιπόν, είναι εμφανής η διασύνδεση στο θέμα των κλιματικών μεταβολών. Η σημερινή πρόκληση σε αυτό το σύστημα ρύθμισης είναι μια αλλαγή στον εξοπλισμό από βραχυπρόθεσμες ερευνητικές δράσεις σε ένα μακροπρόθεσμο και σταθερό πλαίσιο. Το GMS θα μετακινηθεί λοιπόν από την έρευνα και την ανάπτυξη σε δύο επιχειρήσεις. Και αυτή, αυτός είναι ο σκοπός ακριβώς αυτής της ρύθμισης, να δημιουργηθεί δηλαδή μια γέφυρα μεταξύ των προπαρασκευαστικών δράσεων ε, τις οποίες έχετε, για τις οποίες έχετε συμφωνήσει για το 8, 9 και 10 και τις προσεχείς δημοσιονομικές προοπτικές που ξεκινά το 2014. Υπάρχουν ε, δύο έρευνες αξιολόγηση των επιπτώσεων και η ανάλυση των επιπτώσεων προτείνει η Επιτροπή να διασφαλίσει το συντονισμό του GMS και της εφαρμογής του προγράμματος αντί να εκχωρήσει τη λειτουργία αυτή σε έναν ανεξάρτητο φορέα, σε ένα κυβερνητικό φορέα, κυβερνητικό οργανισμό. Δεύτερον, η χρηματοδότηση της Επιτροπής είναι προτιμητέα από, ήπιες, από ήπια μέτρα. Ο ρύθμιση την προτείνει να, υπάρξουν να υπάρξει επιπρόσθετη χρηματοδότηση για την αρχική φάση ε, το 2011, 12 και 13 η χρηματοδότηση που προτείνει η Επιτροπή είναι 150 εκατομμύρια συνολικά. Ο σκοπός αυτής της ρύθμισης καλύπτει ε, την πρόσβαση στα δεδομένα, τις ε, υπηρεσίες όσον αφορά το έδαφος, τους ωκεανούς, την ατμόσφαιρα, τα έκθετα περιστατικά και φαινόμενα κλιματικών μεταβολών. Και εφόσον οι προπαρασκευαστικέ δράσει ολοκληρώνουν το 2010, ε, εξετάζουμε ήδη τις δυνατότητε γεφύρωσης για το 2000, διασύνδεση με το έτος 2011. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Βάισενμπέργκερ. Θα ήθελα να δώσω στον κύριο Γκλάντε τώρα το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Φέσνερ, ευχαριστώ πολύ κύριε Βάισενμπερκ για τις ε, σύντομες και πολύ ξεκάθαρες ε, ε, εισαγωγικές σας παρατηρήσεις. Θα ήθελα όσον αφορά αυτό το σχέδιο κανονισμού το οποίο θα συζητήσουμε να σας πω τα εξής. θα αλλάξουμε όσον αφορά το περιεχόμενο αντίστοιχα όπως το κάναμε για το Γκαλιλαίο. Αλλά δεν θα διαβάσουμε το ίδιο σφάλμα όπως με το Γκαλιλαίο. Αλλά θα, και θα στραφούμε απευθείας προς τη δημόσια χρηματοδότηση. Είναι ενδιαφέρον ότι τα δεδομένα τα οποία θα έχουμε μελλοντικά στη διάθεσή μας θα παρέχονται στις διάφορες υπηρεσίες, φορείς υπηρεσιών στην Ευρώπη δωρεάν και θεωρώ ότι αυτή είναι μια ευκαιρία να συμμετάσχουν νέοι ε, φορείς ε, στην αγορά, να δημιουργούνται με τον τρόπο αυτό νέες υπηρεσίες και να δημιουργούνται νέα μοντέλα, επιστικά μοντέλα. Ε, εντυπωσιακό για μένα συγητή είναι να αναμένω ε, ε, ενδιαφέρον για μένα συγγνώμη να αναμένω τις ε, συζητήσεις που θα ακολουθήσουν ε, της προσεχής με την Επιτροπή Προπολογισμών γιατί το θέμα της χρηματοδότησης είναι ένα ιδιαίτερος ενδιαφέρον πρόγραμμα. Το γνωρίζουμε μάλιστα και από τον Γαλιλαίο όπου πραγματικά υπήρχαν ε, ήταν πολύ δύσκολο να βρεθούν τα κονδύλια. Κατά πόσο τα κονδύλια θα είναι αρκετά, δεν ξέρω, αυτό θα το δούμε. Αλλά θα πρέπει ανεξάρτητα από όλες αυτές τις ε, αμφιβολίες που υπάρχουν ε, είμαι σίγουρος θα δημιουργηθούν πολύ ενδιαφέρουσες υπηρεσίες με τον τρόπο αυτό και θα ήθελα η Κομισιόν να μας πει κάποια πράγματα σε σχέση με τη θέση του Συμβουλίου αν υπάρχουν κάποιες εξελίξεις αν η Προεδρία και τα άλλα μέλη του Συμβουλίου αυτή τη στιγμή είναι πιο ανοιχτά όσον αφορά το θέμα της ε, χρηματοδότησης. Αυτή τη στιγμή ε, βρίσκεται η διαδικασία συνδιαλλαγή σε εξέλιξη με το Συμβούλιο ε, σε σχετικά με τη χρηματοδότηση από το 2014. Επίσης θα ήθελα να σας υπεσχεθώ ότι πραγματικά το χρονοδιάγραμμα είναι ιδιαίτερος, ε, να είναι ιδιαίτερος φιλόδοξο. Ε, κατά πόσο ε, θα υπάρξει συμφωνία στην πρώτη ανάγνωση δεν ξέρω, θα ήθελα να επιφαθώ σχετικά. Τον πρώτο χρόνο είχαμε μια πληθωριστική εξέλιξη, θα έλεγα, στην πρώτη ανάγνωση. Αν δεν υπάρξουν μείζωνα προβλήματα, κατά πάσα πιθανότητα κάτι είναι εφικτό. Αλλά θα ήθελα ευθύ εξ να σας πω ότι θα πρέπει να δούμε ποια είναι η θέση του Συμβουλίου, που υπάρχουν δυνατότητες συμβασμού, ποιες είναι οι αδρές ε, γραμμές ε, συμφωνίας κλπ. Και που μπορούν να υπάρξουν επικοδηματικές ε, προτάσεις. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Επόμενος συνάδελφος, ο κύριος Μπρέζινα. Děkuji za slovo, Eh, Αυτή η έκθεση είναι πάρα πολύ σημαντική, διότι με τα στοιχεία που μπορούμε να πάρουμε από το σύστημα θα μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε σε πάρα πολλούς τομείς από τις ε, ε, θετικές επιστήμες, περιβάλλον, ανάπτυξη των πόλεων κλπ. Θα ήθελα να τονίσω μία ιδιαίτερα εφαρμογή που εγώ τη θεωρώ ιδιαίτερα σημαντική. Η πυροπροστασία. Διότι στο Ευρωκοινοβούλιο σχεδόν κάθε χρόνο συζητάμε πυρκαγιές, ιδιαίτερα στη Νότια Ευρώπη. Και έχουμε ψηφίσει μέτρα αλληλεγγύης. Οι πληροφορίες λοιπόν και το να ξέρουμε γενικά τι συμβαίνει είναι χρήσιμο μόνο όταν τα χρησιμοποιούμε τα στοιχεία αυτά. Κάτι που φαντάζομαι είναι αυτό που σας είπα πριν. Προστασία από τις πυρκαγιές. Γι' αυτό χρειαζόμαστε μία εφαρμογή που να ξεκινάει με το τι γίνεται στο υπερέρυθρο φάσμα και πώς μπορεί να γίνει σωστή διαχείριση όσον αφορά την προστασία. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα. Ευχαριστώ. Πρόεδρος. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μπρετζίνα. Κύριε Τσίζεστε. Um, uh, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Μία γενική παρατήρηση, μάλλον μερικές γενικές παρατηρήσεις καταρχήν. Από την εμπειρία μου από μια αποστολή αντιπροσωπείας ε, της Επιτροπής μας πέρυσι που πήγαμε στην Ρώμη, στην Ίσα, κοντά στη Ρώμη τέλο πάντων. Μια πολύ ενδιαφέρουσα ενημέρωση εκεί για το GMS, e το σύστημα αυτό και άλλα συστήματα ε, που έχουν σχέση με την ραδιοπαρακολούθηση της γης. Ο Σνέφος Γκλάντε αναφέρθηκε στο Γαλιλαίο. Εγώ θα ήθελα να πω ότι το πρόγραμμα αυτό, το GMS, e είναι μια επιτυχία όσον αφορά την πολιτική διαστήματος της Ένωσης. Και θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε να την ενθαρρύνουμε. Και να δείξουμε σε όλο τον κόσμο ότι είναι κάτι πολύτιμο. Θα ήθελα να ακούσω περισσότερα πράγματα για τη λειτουργία του συστήματος, όπως θα λειτουργεί καθοδόν. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Οντί. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ την Κομισιόν που βάζει την Ένωση στο κέντρο ενός σοβαρού προβληματισμού των πολιτών η εξέλιξη της μοίρα του πλανήτη για συλλογή πολύτιμων πληροφοριών για πάρα πολλά όργανα. Ο εισηγητής μας μας είπε ότι οι πληροφορίες αυτές θα είναι δωρεάν θα ήθελα να πάρει θέση από αυτού η Κομισιόν, διότι βγαίνουν χρήματα από τον προπολογισμό της Ένωσης. Δεν θα το έβρισκα παράλογο οι πληροφορίες αυτές να πληρώνονται. Είναι ένα είδος απόδοσης, μιας επένδυσης. Έπειτα, τι θα γίνει με τους μη Ευρωπαίους που θα πάρουν αυτές τις πληροφορίες. Άρα αυτοί που δεν έχουν χρηματοδοτήσει το σύστημα. Έπειτα υπάρχει ένας άλλος κίνδυνος. Η σύγκριση με τον Γαλιλαίο. Το Γαλιλαίο είναι 3 με 4 δις. Δεν είναι στην ίδια κλίμακα. Εδώ μιλάμε για άλλο είδος ποσά. Αν δεν μπορούμε να βρούμε 150 εκατομμύρια για το πρόγραμμα αυτό εδώ, για το οποίο από ό,τι φαίνεται υπάρχει συνένεση πολιτική, αυτό ε, θα δείξει ότι είμαστε ανίκανοι να κάνουμε κοινά προγράμματα. Άρα η σύγκριση με το Γαλιλαίο... Ε, θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί όταν ε, επιχειρούμε να την κάνουμε. Ο κύριος Λάμπερτς. Ευχαριστώ πρόεδρε και συνάδελφοι. Συμφωνώ με πολλά από τα προηγούμενα σχόλια. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο το έχουμε συζητήσει πολλές φορές και μας δίνει την ευκαιρία να συζητήσουμε πολλά θέματα. Η αλλαγή του κλίματος είναι ένα από τα θέματα, αλλά επίσης και η γενική στρατηγική μας, η στρατηγική της ασφάλειας, επάρκειας κλπ πολυδιάστατο θέμα. Δεν θα πρέπει λοιπόν να μας διαφύγει αυτή η ευκαιρία για να, πώς να το πω, πουλήσουμε την δουλειά, την, την αξία που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι εργασίες τις οποίες κάνει στους πολίτες της. Ε, βεβαίως το θέμα εδώ δίδει χρημάτων όπως λένε και πολλών χρημάτων, αλλά αυτό είναι ένα θέμα στο οποίο μπορούμε να προβάλλουμε την αξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους πολίτες της. Γι' αυτό θα πρέπει να ε, φροντίσουμε ε, να μην χρησιμοποιήσουμε τα χρήματα των φορολογουμένων για να κερδοσκοπήσουν ορισμένες εταιρείες. Εντάξει, ε, να χρησιμοποιήσουμε χρήματα των φορολογουμένων εφόσον αυτά επιστραφούν ως αξία δηλαδή των έργων που θα ωφελήσουν τους φορολογούμενους. Θα πρέπει λοιπόν ένα μέρος των κερδών του ωφέλους να εισρεύσει πάλι στις τσέπες των φορολογούμενων. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την υπόδειξη, ιδίω ε, στις περιπτώσεις όπου υπάρχει μεγάλη προστιθέμενη αξία στα μεγάλα έργα για τους, Ευρωπα... για τους Ευρωπαίους πολίτες. και νομίζω ότι πραγματικά αξίζει η συμβολή μας. Η κυρία Ρουσ... Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. <clears throat> Δεν θα μακρηγορήσω. Θα ήθελα μόνο να πω, όπως είπαν και οι συνάδελφοι προηγουμένως, ότι όντως είναι άκρος ενδιαφέρον αυτό το πρόγραμμα για την τηλεπισκόπηση, γεωσκόπηση, για τη διαχείριση των ε, εκτάκτων καταστάσεων, την ασφάλεια, την ατμόσφαιρα, ε, τους ωκεανούς ε, και τα λοιπά και την υπερθέρμανση του πλανήτη. Όλα αυτά ωραία είναι, αλλά εγώ έχω την εξή επιφύλαξη. Μέχρι τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι ηγείτο, δεν είχε το leadership όπως λέμε. Καλό θα είναι λοιπόν να κάνουμε μια προσπάθεια να ανακτήσουμε λίγο βάρος και να βρούμε τη θέση μας σε αυτό το τομέα. Χωρίς να θέλω να το συγκρίνω με το Γαλιλαίο. Θέλω να σας πω το εξή. Όταν είδαμε τι καθυστέρηση έχει τραβήξει ε, το πρόγραμμα Γαλιλαίος. Ε, τώρα ενθουσιαζόμαστε, αλλά τελικά μπορούμε να οδηγηθούμε σε λίγα χρόνια σε αποτελμάτωση, όπως με το Γαλιλαίο. Τι χρειάζεται λοιπόν. Βλέπουμε ότι όλοι έχουμε τη βούληση. Εμείς ναι, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ναι, τα κράτη-μέλη θα χρειαστεί να βάλουν το χέρι στην τσέπη. Εκεί ε, ρωτώ, συμφωνούν όλα τα κράτη-μέλη για αυτό το σχέδιο για να δώσουν συνέχεια. Γιατί εκεί είναι ο φόβος και ανησυχία η δικιά μου. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Βέμπερ ευχαριστώ και εγώ δεν θα μακρηγορήσω. Σύμφωνα με αυτά που μας είπε η Κομισιόν και αντίθετα με τις απόψεις συναδέλφων που μίλησαν, εγώ επιμένω στη σημασία της ελεύθερης πρόσβασης και του δωρεάν χαρακτήρα των πληροφοριών. Διότι στην υπόθεση αυτή έχει σημασία όχι να δούμε μόνο τους δορυφόρους, το hardcore όπως το λέμε, αλλά να αναπτυχθεί και η αγορά υπηρεσιών, να πολλαπλασιάσουμε τους χρήστες. Θα ήταν τραγικό για μια φορά ακόμη να φτιάξουμε μια υποδομή, να φτιάξουμε τους δορυφόρους, που πρέπει να συμπληρωθούν βέβαια και αυτό είναι ένα ερώτημα που το θέτω, γιατί σήμερα έχουμε πέντε δορυφόρους παρατήρησης. Πώς σκοπεύουμε να συνεργαστούμε με τους Αμερικάνους, τους Ιαπωνέζους, τους Ινδούς που έχουν άλλους δορυφόρους γιατί για μια σοβαρή γεωεπισκόπηση δεν αρκούν πέντε δορυφόροι, χρειάζονται 30 δορυφόροι και θα χρειαστεί χρόνος για να γίνουν όλα αυτά. Χρειάζεται λοιπόν συνέργεια μεταξύ των δορυφόρων του δικού μας συστήματος και των δορυφόρων των άλλων συστημάτων πρέπει να οργανωθεί. Βέβαια υπάρχουν όργανα στη Γενέβη που ασχολούνται με αυτά και επανέρχομαι και πάλι στην ανάγκη να δημιουργηθεί η αγορά. Οι ασφαλιστές, οι χρήστες, οι οι χρήστες των πληροφοριών. Ελεύθερη πρόσβαση δωρεάν. Αυτό πρέπει να διασφαλιστεί. Ευχαριστώ πολύ ο κύριος Αντιπρόεδρος Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να προσθέσω κάτι εν συντομία. Πολλοί ε, συνάδελφοι είχαν θετική άποψη από αυτού του θέματος και πιστεύω ότι εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορέσει να προβάλλει αξιόπιστα στοιχεία και επιβεβαιωμένα στοιχεία, στοιχεία για έναν μεγάλο αριθμό χρηστών στις αστικές περιοχές, στις ε, διάφορες, ε, ε, στα διάφορα κράτη και στις γεωγραφικές περιοχές. Αυτό θα αποδειχθεί πάρα πολύ χρήσιμο για να υπερασπίσουμε την αντικειμενικότητα των στοιχείων αυτών. Εγώ δεν είμαι ειδικό ε, στην στατιστική και στην έρευνα, αλλά πιστεύω ότι θα πρέπει τα στοιχεία αυτά να βασίζονται όσο το δυνατόν μεγαλύτερο αριθμό ε, μεγαλύτερων περιοχών και γεωγραφικών εκτάσεων για να είναι ε, αξιόπιστα. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε αντικειμενικοί και αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό στοιχείο η αντικειμενικότητα και η αξιοπιστία των στοιχείων. Ε, δεν μπορούμε σήμερα να φανταστούμε τις, ε, όλες τις ε, πιθανές χρήσεις αυτής της τεχνολογίας, όλο το φάσμα το οποίο θα αναπτυχθεί βάσει αυτού του συστήματος. Μόνο όταν το σύστημα αυτό εφαρμοστεί και δοκιμαστεί θα μπορέσουμε να κατανοήσουμε όλο το εύρος και όλες τις δυνατότητες που προσφέρουν αυτά τα στοιχεία τις δύο σκόψεις. Πιστεύω ότι εδώ παρουσιάζεται μια θαυμάσια ευκαιρία για την Ευρωπαϊκή Ένωση να δράσει. Κάποιος είπε ότι δεν βλάπτει να κάνουμε μια ανασκόπηση της δύσκολης, της περίπλοκης ιστορίας, του περίπλοκου παρελθόντος του Γαλιλαίου. Συμφωνώ καλό είναι να θυμηθούμε, να μελετήσουμε το παρελθόν του Γαλιλαίου και του συστήματος για να αποφύγουμε ε, παρόμοια λάθη στο μέλλον. Ξέρουμε ότι όλη αυτή βεβαίω η άσκηση θα είναι πανάκριβη, διότι δορυφορικά στοιχεία είναι τα πιο ακριβά στοιχεία, τα οποία ε, παρέχονται και Αυτό που επίσης πρέπει να φροντίσουμε είναι τα στοιχεία αυτά να παραμείνουν διαφανή, να είναι καθαρά στοιχεία, όχι αλλοιωμένα και ε, να διατεθούν όσο το δυνατόν νωρίτερα. Έτσι θα μπορέσουμε να μειώσουμε την απόσταση μεταξύ πολιτών και Ευρωπαϊκής Ένωσης το οποίο δεν μπορεί να γίνει μόνο από την, τα κράτη-μέλη. Η προστιθέμενη αξία δηλαδή μεγάλη. Ε, η κυρία Χόρ Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να σχολιάσω σύντομα τα σχόλια τα οποία έγιναν για την καταβολή του κόστους, το πόσο θα πληρώνουμε και αν ε, θα πρέπει οι δημόσιες αρχές να έχουν ελεύθερη πρόσβαση, δηλαδή δωρεάν πρόσβαση στα στοιχεία ή όχι και πώς θα γίνεται η καταβολή του τιμήματος αν υπάρχει. Νομίζω ότι υπάρχει μεγάλη προστιθέμενη αξία και υπάρχουν χώρες που ήδη έχουν ε, ε, εφαρμόσει αυτό το σύστημα σε χώρες της Αφρικής, παραδείγματος χάρη, για να παρατηρήσουν ε, την ε, παρατήρηση στην δασοπονία, συντήρηση δασών κλπ. Ε, όσον αφορά τις προσαρμογές, θα πρέπει να μελετήσουμε προσεκτικά τι δεσμεύσεις θα αναλάβουμε και τι θα προσφέρουμε. Παραδείγματο χάρη μπορούμε να προσφέρουμε μέσω του συστήματος αυτού στις χώρες που υποφέρουν να παρέχονται συγκεκριμένε πληροφορίες που θα τις βοηθήσουν να ανταπεξέλθουν στις δυσκολίες τους. Είμαι λοιπόν πολύ επιφυλακτική όσον αφορά τον περιορισμό της πρόσβασης σε αυτά τα στοιχεία. Και πιστεύω ότι από τη δική μας πλευρά πρέπει να παίξουμε ένα σημαντικό ρόλο στην προσαρμογή του συστήματος και τη χρήση του σε δύσκολες περιοχές του κόσμου. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Ντατή. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε για την πρόταση για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Γεωσκόπησης που ενέκρινε η Κομισιόν πέρυσι. Χαίρομαι ιδιαίτερα για το ότι η ομάδα ΕΛΚ με όρισε σκιώδη συγγήτρια για την λειτουργική λοιπόν ικανότητα παρατήρηση τη γης η Ένωση με έναν διαρκή τρόπο εξασφαλίζει στα μέσα να αντιμετωπίσει νέε προκλήσει και όσον αφορά την αλλαγή του κλίματο, και τη διαχείριση των φυσικών πόρων και την ασφάλεια των συμπολιτών μας. Το βλέπουμε αυτό στην επικαιρότητα. Δεν τι έγινε το Σαββατοκύριακο. Θλιβερά ξαναθυμηθήκαμε την ανάγκη να πρόληψης φυσικών καταστροφών και θερμινιών. Το είδαμε στην Μανίλα με τις πλημμύρες, χειρότερες πλημμύρες των τελευταίων 40 ετών που νομίζω είχαν πάνω από 140 θύματα ένα θλιβερό παράδειγμα μεταξύ άλλων αποδεικνύει την ανάγκη και τον επίγοντα χαρακτήρα εφαρμογής ενός τέτοιου προγράμματος για καλύτερη προ... πρόβλεψη, πρόληψη μάλλον των κινδύνων. Βέβαια πρέπει δούμε την αξιολόγηση των δημοσίων πολιτικών και στη συγκεκριμένη περίπτωση η διαχείριση σε θέματα χωροταξίας παραδείγματος χάρη. Το πρόγραμμα αυτό θα μας δώσει τη δυνατότητα για μια πιο εύστοχη ε, διαχείριση σε θέματα χωροταξία. Επίσης, θα επιτρέψει να αντιμετωπιστούν ε, προκλήσεις όπως ε, στην Κοπεχάγη που συσχέτει το θέμα της πυρκαγιάς των δασών, υπερβολικής αστικοποίησης. Και στο σημείο αυτό έρχομαι σε αυτά που είπε ο κύριος Βέμπερ πριν, δηλαδή ο ιδιωτικό τομέας θα πρέπει να έχει πρόσβαση στις πληροφορίε αυτές και αυτό θα αυξήσει και την παραγωγικότητα. Παραδείγματο χάρη σε μια εταιρεία παραγωγή πετρελαίου θα μπορεί να κρίνει πού να τοποθετήσει για πιο επικεδή τρόπο μια πλατφόρμα στη θάλασσα για το πετρέλαιο. Επίση, στι ε, νέε τεχνολογίε για τη γεωργία και που συνδέονται και με την διαρκή αένα ή ανάπτυξη. Ή αν έχουν οι επιχειρήσεις πρόσβαση σε αυτά τα στοιχεία θα τους είναι χρήσιμο. Και τώρα έχουμε σε τρεις ερωτήσεις μια τεχνική διαφοροποίηση των πηγών χρηματοδότησης. Με χρηματοδότηση από το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο και ειδική χρηματοδότηση στην εφαρμογή αυτού του κανονισμού είναι δύσκολο και για μας και για αυτούς που μας εξέλιξαν να παρακολουθούμε όλες τις συνιστώσεις, πώς θα χρηματοδοθούν μόνο όλες τις συνιστώσεις. Να οριστούν λοιπόν οι πηγές χρηματοδότησης και το ποσό για κάθε πηγή. Δεύτερη ερώτηση. Η σωστή διακυβέρνηση του προγράμματος. Είχαμε μια ανακοίνωση πρόσφατη σχετικά με το πρόγραμμα και αναφέρεται ένα συμβούλιο εταίρων. Κονσέγγιντε παρτένερ. Αυτοί οι εταίροι τι καθεστώς έχουν. Από τι θα απαρτίζει το Συμβούλιο από εκπροσώπου των κρατών μελών που συμβάλλουν στο πρόγραμμα αυτό για την υποδομή. Πάντως, οπωσδήποτε το Συμβούλιο αυτό και οι εταίροι θα έπρεπε να έχουν μόνιμα μέλη προκειμένου να πετύχει το πρόγραμμα αυτό. Το ίδιο ισχύει και για τη χρηματοδότηση. Όσο πιο σαφεί είμαστε για τη χρηματοδότηση και για τα σχετικά κριτήρια, τόσο το καλύτερο. Το ίδιο και για τη χρηστή διαχείριση. Τέλος, η μελλοντική εξέλιξη του προγράμματο. Για την καλή λειτουργία του προγράμματο πρέπει να έχουμε αποτελεσματική συνεργασία με τις αξίες της Κομισιόν και των κυβερνήσεων. Καλό είναι να υπάρχει αυτό το Συμβούλιο, αλλά και η σύνθεση θα πρέπει να την ξέρουμε και το καθεστώς που θα ισχύει. Η πρόταση κανονισμού δεν αναφέρεται πουθενά στο Συμβούλιο αυτό εταίρων. Έπειτα, αν γίνει αυτό το Συμβούλιο εταίρων, ή είναι στην ημερήσια διάταξη, με τι προθεσμίες, πότε σκοπεύει να προβεί στη σύνθεση αυτού η Κομισιόν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα δεν έχει ζητήσει κανένα άλλο συνάδελφο το λόγο. Θα παρακαλούσα τον κύριο Βάισεμπερκ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να απαντήσει. Πολλέ οι ερωτήσει που σα έγιναν. Μήπω θα μπορούσατε να απαντήσετε σε ορισμένε ή σε πολλέ. Κατά τα άλλα, υποθέτω ότι θα δοθεί και συνέχεια στι ερωτήσει, αν δεν μπορείτε να τι απαντήσετε τώρα. Ήταν σημαντικέ ερωτήσει που αφορούν λεπτομέρειε όμω. Έχετε το λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχάς, πώς έχει η κατάσταση στο Συμβούλιο. Έξι συμβούλια για την ε, διάστημα έγιναν μέχρι τώρα και σε όλα αυτά τα συμβούλια συζητήθηκε το σύστημα GMES και οι αρμόδιοι υπουργοί είπαν ότι όλα αυτά τα οποία έχουμε επενδύσει για την έρευνα και ανάπτυξη θα πρέπει εκ των υστέρων να εισέλθει, να ενσωματωθεί στην επιχειρησιακή, στον επιχειρησιακό τομέα. Η συγκεκριμένη πρόταση λοιπόν παρουσιάστηκε πριν από μερικές μέρες στο Συμβούλιο ακριβώς όπως σας την παρουσίασα εγώ και οι διαβουλεύσεις στο Συμβούλιο θα αρχίσουν Τώρα η πολιτική βούληση του Συμβουλίου Υπουργών Αρμοδίων για το διάστημα το έχει επιβεβαιώσει ότι επισημεί το σύστημα αυτό. Ε, οι Υπουργοί έχουν επίσης επιβεβαιώσει ότι επισημούν την ελεύθερη πρόσβαση στα, στα στοιχεία αυτά. Από την έρευνα που έχουμε κάνει έχουμε διαπιστώσει ότι τα ε, ε, συστήματα τα οποία έχουν ε, κατιούσα πορεία λειτουργούν καλύτερα όταν η είσοδος και η χρήση των στοιχείων αυτών είναι ελεύθερη. Πέραν αυτού, οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, το Emergency Services ή το GMES, είναι μία από τις υπηρεσίες οι οποίες έχει αγκριθεί στην προπαρασκευαστική βάση, στην προπαρασκευαστική φάση από εσά και συζητείτε αυτή τη στιγμή. Η διάθεση του κεφαλαίων για το GMES για έκτακτες ε, ανάγκες ε, και επεμβάσεις ε, η μη στρατιωτικής φύσεως είναι απαραίτητη και έχουμε θέσει ένα πιστώσεις για αυτό το σκοπό επεμβάσεις περίπτωση πυρκαγιάς και χρήση του συστήματος για έκτακτες ανάγκες. Ε, αυτή τη στιγμή αναπτύσσεται μια πρωτοβουλία πολιτών για την παρακολούθηση του συστήματος η οποία δεν λειτουργεί απομονωμένα αλλά σε παγκόσμια, παγκοσμίως υπάρχει ε, μία, ένα σύστημα που λέγεται ε, GESS Global ε, Observation System of Systems δηλαδή είναι ένα σύστημα γεωσκόπησης το οποίο χρησιμοποιείται από τους Κινέζους, τους Ινδούς, τους Αμερικανούς από όλα τα μέρη του κόσμου και το οποίο διαθέτει τα συλλεγόμενα στοιχεία δωρεάν Εάν λοιπόν εμείς διαθέσουμε τα στοιχεία μας ε, ελεύθερα, δωρεάν, θα έχουμε και εμείς ελεύθερη πρόσβαση σε αυτό το παγκόσμιο γεωσκοπικό σύστημα, παγκόσμιο σύστημα γεωσκόπησης. Όσον αφορά την παρατήρηση της κυρίας Ντατή, η οποία ρώτησε αν θα πρέπει τώρα να ε, προβάλλουμε την πρόταση αυτή, να περιμένουμε μέχρι την επόμενη ε, χρηματοδοτική περίοδο, δημοσιονομική περίοδο, ε, απαντώ ότι αποφασίσαμε να το προωθήσουμε τώρα για να μην χαθούν ορισμένες ερευνητικές πτυχές και χάσουν τη χρηματοδότησή τους οι οποίες χρειάζονται για το GMES το εν συνεχεία το 2012-2013 θα πρέπει οπωσδήποτε να φροντίσουμε για την κάλυψη των, ε, ε, των πιστώσεων που χρειάζονται. Γι' αυτό ακριβώς αυτό το μεσοδιάστημα από σήμερα μέχρι το 2012-2013 είναι ε, ένα, μια περίοδος γεφύρωσης για την μελέτη επιπτώσεων την οποία έχουμε κάνει, έχουμε συντάξει δείχνουν ότι εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση προχωρήσει και αποκτήσει τα στοιχεία ή αγοράσει τα στοιχεία για το GMES, τότε το κόστος των αποκτησέντων στοιχείων ε, μειώνεται και δημιουργείται μια καλύτερη σχέση κόστους-οφέλους. Ε, όσον αφορά τώρα την Αφρική, εδώ και δύο χρόνια έχει αναπτυχθεί μια πρωτοβουλία από τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ένωσης Αφρικαϊκών Κρατών ε, ένα έργο δηλαδή το οποίο θα ε, στοχεύσει αποκλειστικά στην ανάπτυξη της Αφρικής και πάλι τα στοιχεία αυτά τα οποία θα διατίθενται ε, στην Αφρική, ε, στους χρήστες από την Αφρική είναι δωρεάν και εντάσσεται και στα πλαίσια της αναπτυξιακής βοήθειας αλλά και της προστασίας του κλίματος. Τώρα, για την Κοπενχάγη σκεφτόμαστε μήπως θα μπορέσαμε μέσα σε αυτό το πλαίσιο να ε, εισαγάγουμε και ένα στοιχείο αλλαγής του κλίματος ε, διότι ε, ενδέχεται σε όλο το φάσμα των συζητήσεων για την αλλαγή του κλίματος να δημιουργηθεί μια απόκληση. Ίσως μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε και αυτό το στοιχείο. Τώρα, η πηγή της χρηματοδότησης. Μέχρι τώρα το EMS χρηματοδοτήστηκε αποκλειστικά από το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα και την ανάπτυξη και ορισμένα στοιχεία του όπως η λειτουργία δορυφόρων, δορυφόρων το 2012 δεν έχει πλέον καμία σχέση με την έρευνα. Και γι' αυτό θα πρέπει το πλαίσιο να, να, να εγκαταλείψουμε, να βγούμε εκτός πλαισίου ε, ερευνητικής ε, υποστήριξης και να το εντάξουμε σε ένα νέο πρόγραμμα, σε ένα νέο πλαίσιο. Έχουμε λοιπόν ακριβώς ένα νέο πλαίσιο τον θα δημιουργήσουμε για να εντάξουμε το GMES. Όσον αφορά την πρόταση αυτή τα 150 εκατομμύρια, είναι ένα μείγμα από την αναδιάρθρωση της ανάπτυξης του τίτλου Α και τη χρησιμοποίηση των υπολείπων εκατομμυρίων κατά διαφορετικό τρόπο ε, σε συνδυασμό με το υπόλοιπο από την έρευνα και τεχνολογία. Μία λοιπόν αναδιάρθρωση των κονδυλίων. Η... Πώς θα διαμορφώσουμε τώρα τις σχέσεις μας με τα συμμετέχοντα κράτη, με τα κράτη-μέλη. Ε, αντίθετα από ό,τι στο, είχε γίνει στο πρόγραμμα Γαλιλαίος, το GMES είναι ένα ε, πρόγραμμα συνεργασίας, ένα, ένα έργο συνεργασίας και αυτή η συνεργασία θα πρέπει να διαπεράσει όλα τα αρμόδια όργανα και όλους τους, ε, τα σεισμικά όργανα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Πιστεύω ότι ήταν μια εμπεριστατωμένη ε, απάντηση αυτή. Ε, αναφερθήκατε συγκεκριμένα στις διάφορες πτυχές και θα ήθελα ε, κατακλείδω να δώσω το λόγο στον κύριο Γκλάντε, στον εισηγητή. Ευχαριστώ πολύ σύντομα. Σας έχω πει ότι υποστηρίζω το, το πρόγραμμα αυτό και χαίρομαι πολύ που περιοριζόμαστε στα ουσιαστικά σημεία διότι ο χρόνος είναι χρήμα και γι' αυτό ήμουν και έτσι τηλεγραφικός. Από ό,τι κατάλαβα, το, υπάρχουν ορισμένες επιφυλάξεις από συναδέλφους ε, και ε, επειδή ε, εάν υπάρχουν ερευνητικά αποτελέσματα τότε θα πρέπει τα συμπράσματα αυτά να ενσωματωθούν στην ανάπτυξη διαφορετικά τι να τα κάνουμε, τι να κάνουμε την έρευνα δεν ξέρω αν είναι κατάλληλη στιγμή τώρα να μιλήσουμε για το χρονοδιάγραμμα, αλλά θα έλεγα να είμαστε προσεκτικοί, να μην είμαστε υπερβολικά φιλόδοξοι. Το Δεκέμβρη να υποβληθεί η έκθεση και ε, να κάνουμε τις ε, συζητήσεις επ' αυτής. Και εάν οι συνάδελφοι συμφωνούν, θα είμαι, πρόθυμο είμαι πρόθυμος να την διαμορφώσω την έκθεση αυτή μέχρι το Δεκέμβρη και να αρχίσουμε τις συζητήσεις. Ευχαριστώ κύριε Γκλάντε. Ακόμα δεν έχουμε ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, δεν έχουμε πρόταση, αλλά θα παρακαλούσα και τους συναδέλφους να προχωρήσουν ε, γρήγορα. Είναι πάρα πολλά θέματα στη διαδικασία διαβούλευσης και ε, ε, όσο μπορούμε ταχύτερο καλό είναι να ξεκινήσουμε τη συζήτηση για το θέμα αυτό γιατί δεν πιστεύω ότι υπάρχει κάποια μεγάλη διαφωνία ή αμφισβήτηση του, του θέματος αυτού. Ο εισηγητής ε, προτείνω ε, τη δεύτερη εβδομάδα του Οκτωβρίου 12 με 15 ίσως να παρουσιάσω την ε, έκθεση με, τα, με ενσωματωμένα τα σχόλια και τις παρατηρήσεις των συναδέλφων που ακούστηκαν σήμερα Ωραία, πολύ ωραία, λέει ο πρόεδρος, θερμά ευχαριστώ και ολοκληρώσουμε αυτό το σημείο, εάν δεν επισημεί κάποιος το λόγο, ωραία, και προχωρούμε στο 4. Δομές διαχείρισης για τα ευρωπαϊκά προγράμματα δορυφορικής ραδιοπλοήγησης. Έχετε την πρόταση και λέω να συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο, να δώσουμε το λόγο στον εκπρόσωπο της Κομισιόν. Καταρχάς, ο κύριος Πάουλ Φέρχοφ. Σας δίνω το λόγο και να μας κάνετε μια σύντομη παρουσίαση. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Λέω Αλμαν Χοφ. Είμαι υπεύθυνος για το θέμα αυτό της δορυφορικής ραδιοπλοήγησης και θα συνεργαστώ με την Επιτροπή σας στη νέα της Πριν όμως πω δύο λόγια για την πρότασή μας για τον κανονισμό αυτό. Αξίζει να δούμε μερικά στοιχεία σχετικά με το που βρισκόμαστε στην αφορά το Νομίζω ότι αυτό ενδιαφέρει πολύ την Επιτροπή σας. Και ας τα πω από την αρχή τους, ώστε να μην γίνονται ερωτήσεις από αυτόν αργότερα. Την 1η Οκτωβρίου, δηλαδή σε λίγες μέρες, σκοπεύουμε να κλείσουμε τα συμβόλαια για την λειτουργία από την 1η Οκτωβρίου μέχρι το τέλος του 2013 η ανοιχτή υπηρεσία του Άγνος λοιπόν θα αρχίσει να λειτουργεί από την 1η Οκτωβρίου. Το ανακοινώνουμε αυτό επίσημα και μέσω του τύπου Αξίζει να σημειωθεί αυτό το στοιχείο ότι τέλος ορίμασε η κατάσταση και είμαστε σε θέση να έχουμε αυτή την υποδομή δορυφορικής ραδιοπλοήγησης. Για το Καγγελαίο έχουμε δύο δορυφόρους, όπως ξέρετε, οι οποίοι λειτουργούν. Είμαστε στη φάση τροχιάς αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν συγκεκριμένα σημεία στον κόσμο που είναι εξοπλισμένα όπου κατασκευάζονται οι δορυφόροι και ο στόχος είναι οι δύο πρώτοι δορυφόροι να εκτοξευθούν τον Νοέμβριο του 2010 και οι άλλοι δύο στις αρχές του 2011. Για το αυτό που λέμε FOC, πλήρη λειτουργική ικανότητα του Γαλιλαίου, με τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας για το διάστημα, γίνονται οι αγορές, οι προμήθειες, που, όπου προβλέπετε ότι έξι μεγάλα πακέτα θα αγοραστούν από το βιομηχανικό κλάδο, υποστήριξη συστημάτων, δύο συμβόλαια για την υποδομή εδάφους, ένα συμβόλαιο για τους ε, εκτοξευτές, ένα για τους δορυφόρους και ένα για τη λειτουργία. Προβλέπουμε αυτή τη στιγμή να δοθούν τρία συμβόλαια για τρία από τα πακέτα αυτά μέχρι το τέλος του χρόνου. Υποστήριξη συστημάτων το ένα, δορυφόροι το δεύτερο και ενδεχομένω και εκτοξευτές. Τον να υπάρχουν οι πιο καλές προσφορές, αυτό θα το μελετήσουμε τις επόμενες εβδομάδες. Από ό,τι βλέπω έχετε προχωρήσει κι εσείς στις πολύπλοκες διαπραγματεύσεις με τη βιομηχανία για το θέμα αυτό, όπως θα έχετε διαπιστώσει. Παράλληλα, έχουμε και προτάσεις προς εσάς και προς το Συμβούλιο για τις αρχές του επόμενου χρόνου, ως προς το πώς θα εφαρμοστούν τα προγράμματα μετά το 2013, διότι όπως ξέρετε ο προπολογισμός φτάνει μέχρι τότε. Πρέπει να οργανώσουμε και την μακρόπνοη χρηματοδότηση και την διαχείριση των προγραμμάτων μακροπρόθεσμα με προτάσεις μας. Η πρόταση δεν θα αφορά μόνο την επόμενη δημοσιονομική περίοδο. Οι προτάσεις θα αφορούν και το πώς θα γίνονται οι προμήθειες, η ανάπτυξη, η λειτουργία ενός τέτοιου συστήματος για τις επόμενες δεκαετίες. Τώρα έχουμε στη συγκεκριμένη πρόταση. Θα θυμόσαστε το GSA, δηλαδή η υπηρεσία μας, συναισθήθη από το Συμβούλιο τον Ιούλιο του 2004. Μόλις τότε ξεκινούσε ο Γαλιλαίος με τα πρώτα συμβόλαια. Το PPP ήταν ο, θα ήταν ο φορέας πρώτης λειτουργίας του συστήματος και το δικό μας όργανο ήταν αρμόδιο να ολοκληρώσει τα συμβόλαια και την πρώτη εφαρμογή των προγραμμάτων. Στο τέλος του 2006 η Κομισιόν κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το PPP δεν λειτουργεί σωστά και το 2007 έκανε προτάσεις για πλήρη αλλαγή κατεύθυνσης των προγραμμάτων. Οπότε και ο δικός μας ρόλος του GSA μοιραία έπρεπε να αλλάξει με βάση τη νέα πραγματικότητα. Το 2008 το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο συμφώνησαν για τον κανονισμό 683 ο οποίος στο ρυθμιστικό του μηχανισμό προβλέπει όλους τους κανόνες και μηχανισμούς που χρειάζονται για να λειτουργεί το σύστημα με τη νέα μορφή του. Το υπόλοιπο ήταν επιπλέον προσαρμογές στο έργο του GSA που είναι στον κανονισμό 1321 έτσι ώστε ο κανονισμός 1321 και αυτός να συμφωνεί με τις νέες πραγματικότητες. Η πρόταση λοιπόν που έχετε στα χέρια σας κάνει ακριβώς αυτό. Δηλαδή, εμπεριέχει τα στοιχεία του 1321 ώστε να ευθυγραμμιστεί με τον 683 παραμένει ο στόχος και το όνομα του δικού μας δικής μας υπηρεσίας GSA αυξάνει ο ρόλος της Κομισιόν μέσα στην υπηρεσία αυτή έτσι ώστε η υπηρεσία να αποδίδει το έργο σεβόμενη το ρόλο της Κομισιόν ως διαχειριστή του προγράμματος και ταυτόχρονα μπαίνει και το πλαίσιο ευθυνών της υπηρεσίας προκειμένου να παρέχεται ασφάλεια και οι αναγκαίες εγκρίσεις. Τα κύρια χαρακτηριστικά αυτής της πρότασης είναι ότι περιορίζεται το έργο του, της υπηρεσίας με βάση τα 683, οπότε επειδή ορισμένες αρμοδιότητες περνάνε στην Κομισιόν, αυτό έχει γίνει ήδη εξάλλου, προτίθεται νέο όνομα για την υπηρεσία αυτή, γιατί πρέπει να προσαρμοστεί στο νέο ρόλο της. Διαφορετική διαχείριση του προγράμματος, γιατί όπως σας είπα η Κομισιόν είναι ο διαχειριστής του προγράμματος και σύντομα θα εκδώσει κατευθυντήρες γραμμές προς το GSA, προς εμά δηλαδή. Εμείς θα φροντίσουμε τα προγράμματα να ε, λειτουργούν εγκαίρως. Το 50% των ψήφων τα έχει η Κομισιόν και το εκτελεστικό όργανο της υπηρεσίας θα ασκεί το έργο με βάση τις κατευθυντήρες γραμμές που θα εκδώσει η Κομισιόν. Δεν είναι επομένως απολύτως ανεξάρτητο πια. Επίσης προτείνουμε τη συμμετοχή ως παρατηρητών εκπροσώπων του Κοινοβουλίου στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και το Διοικητικό Συμβούλιο θα έχει λίγο πιο αυξημένο ρόλο στη διαχείριση των της υπηρεσίας, έτσι ώστε η υπηρεσία, το agency, να φέρει σε πέρα στο έργο του όπως έχει οριστεί. Τώρα σχετικά με την αναγνώριση ε, αρμοδιοτήτων και ασφάλειας, security accreditation. Για ένα δημόσιο πρόγραμμα όπως το Γαλιλαίο, το θέμα αυτό της ε, ασφάλειας και της έγκρισης είναι από την εμπειρία μας περισσότερο εθνικό αλλά στη συγκεκριμένη αυτή περίπτωση ε, κοινωνικού προγράμματος πρέπει να υπάρχει και αυτή η συνιστόσα. Πολύ λίγοι εμπειρογνώμονε υπάρχουν στην Ένωση, ιδιαίτερα στις εθνικές διοικησει που να καταλαβαίνουν το έργο αυτό, τη σημασία του και που να μπορούν να το εκτελέσουν. Όπως θα ξέρετε, το έργο αυτό της αναγνώρισης ευθύνης, έγκρισης ευθύνης, έχει σχέση με την ασφάλεια, τις απαιτήσει ασφάλειας και μέσω της διαδικασίας αυτής καλύπτονται οι εθνικοί κίνδυνοι που εμπεριέχονται στο σύστημα. Βέβαια ο κίνδυνος ασφάλειας θα πρέπει να σταθμίζεται ε, με βάση άλλα στοιχεία του προγράμματος. Είναι κάτι το πολύ πολύπλοκο δηλαδή. Εμείς τις προτάσεις μας τις κάναμε με βάση τέσσερις βασικές αρχές. Το έργο θα γίνεται συλλογικά. Θα περιμένουν όλοι οι εμπειρογνώμονες σε θέματα ασφάλειας κλπ. Δεύτερον, θα υπάρχουν οι επιμέρους αποφάσεις Τη Εθνικής Διοίκησης προκειμένου να δοθεί η έγκριση για μια εγκατάσταση είτε για το Γαλιλαίο είτε για την κατασκευή σε ένα εργοστάσιο στο συγκεκριμένο κράτος μέλος αν αυτό είχε επίπτωση στην εθνική ασφάλεια και για κάποιο άλλο κράτος μέλος. Γι' αυτό μιλάμε για την συλλογική ευθύνη. Η επόμενη αρχή θα υπάρχει μια διαρκής διαδικασία εποπτείας όσον αφορά τις εγκρίσεις. Στο σημείο αυτό η υπηρεσία θα παίζει σημαντικό συντονιστικό ρόλο. Η άλλη αρχή είναι η, ότι οι εγκρίσεις αυτές θα εγκρίνονται από επαγγελματίες και οι αποφάσεις θα λαμβάνονται ανεξάρτητα από την Κομισιόν και από τους φορείς που θα είναι υπεύθυνοι για την εφαρμογή των προγραμμάτων και τη λειτουργία του συστήματος. Τέλος, προτείνουμε να υπάρχει και ένας τρίτος πυλώνας στο GSA, πέρα από τον εκτελεστικό διευθυντή δηλαδή και το διοικητικό συμβούλιο, προτείνουμε να υπάρχει μια επιτροπή όσον αφορά την έγκριση σε θέματα ασφαλείας, accreditation, με βάση συμβουλή των εμπειρογνωμόνων. Συνοψίζω. Τι σημασία έχει η πρόταση αυτή για το Κοινοβούλιο. Πρώτον, συνεχίζει την απόφαση που είχε ληφθεί για τα προγράμματα δορυφορικής αδειοπλοήγησης. Να υπάρχει πλήρης ακολουθία μεταξύ των διαφόρων ρυθμιστικών οργάνων και συστημάτων που έχουν εφαρμοστεί τώρα. Δεύτερον, αυξημένος ο ρόλος του Κοινοβουλίου ΕΦΕΞΗΣ. Γι' αυτό πήραμε το άρθρο 156 ως νομική βάση Έπειτα δίνεται και ρόλος παρατηρητή στο Διοικητικό Συμβούλιο, στο Ευρωκοινοβούλιο. Η πρώτη λαμβάνει υπόψη όλα τα αιτήματα του Κοινοβουλίου σχετικά με τις διάφορες υπηρεσίες, δηλαδή βελτιωμένη διαχείριση, δικαιώματα ψήφου για την Κομισιόν, παρακολούθηση της δραστηριότητας των υπηρεσιών, με πλήρη ακολουθία με ευθύνη της Κομισιόν. Επίσης, σεβόμαστε και τους δημοσιονομικούς περιορισμούς προβλήμα αύξηση για το προσωπικό μόνο σε τομείς όπου έχουμε την κύρια ευθύνη στο μέλλον. Δηλαδή δραστηριότητες που έχουν σχέση με την ασφάλεια και όσον αφορά το κέντρο εποπτείας ασφάλειας του Γαλιλαίου. Κύριε Πρόεδρε, με μεγάλη μας ευχαρίστηση, αν γίνεται να υπάρξει πρώτη, σε πρώτη ανάγνωση συμφωνία μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου γιατί για ένα τέτοιο λειτουργικό πρόγραμμα είναι χρήσιμο να έχουμε τα εργαλεία σαφή και έγκαιρα λειτουργικά. Και θα σας βοηθήσουμε και εσάς και τον εισηγητή σας στο έργο σας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για την παρουσίασή σας. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στον εισηγητή, τον κύριο Τοσνόφσκι. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Είμαι πολύ ευτυχής και είναι μεγάλη μου τιμή ως νέο μέλος του σώματος για το γεγονός ότι είμαι συγητής σε έναν τομέα ο οποίος ε, πρόσκειται στην, ε, ε, πολύ, είναι πολύ κοντά με την παλιά μου δουλειά ως μαθηματικού και επιστήμονα. Είναι το έργο αυτό της στάθμης για την Ευρώπη και Γι' αυτό πρέπει να το υποστηρίξουμε με όλες μας τις δυνάμεις. Χαίρομαι που η Κομισιόν θέλει να διευκρινίσει τη διαδικασία λήψης αποφάσεων σε αυτό το λίαν περίπλοκο θέμα, όχι μόνο από τεχνικής πλευράς, αλλά θέλει να διευκρινίσει και όλα τα, τις πτυχές ε, ασφάλειας, ε, χρηματοδότησης ε, και όλων των άλλων πτυχών που εμπλέκονται σε αυτό το έργο. όλες οι συζητήσεις που είχαν γίνει παλαιότερα για τον Γαλιλαίο ήταν πάρα πολύ περίπλοκες και αποφασίστηκε να εγκαταλειφθεί το μοντέλο PPP. Για να βοηθήσουμε το Γαλιλαίο να ε, λειτουργήσει ε, πλήρως. Η πρόταση την οποία έχουμε σήμερα μπροστά μας είναι τεχνικής φύσεως και ορίζει τις ε, αρμοδιότητες της Κομισιόν. Ε, μία συζήτηση, η συζήτηση που θα κάνουμε δεν θα είναι εύκολη, αλλά η πορεία την οποία ακολουθούμε πιστεύω ότι είναι η σωστή πορεία. Ε, θα είναι δύσκολο να αποφασίσουμε για όλες τις τεχνικές και χρηματοδοτικές παραμέτρους ε, ε, στα χρόνια που έρχονται, στο μέλλον, αλλά είναι πολύ σωστή η προσπάθεια της Κομισιόν να καθορίσει ποιος έχει ποιες αρμοδιότητες και να βελτιώσει ε, τον έλεγχο του σώμα του Κοινοβουλίου για τη ροή των κονδυλίων. Αυτό που θα είναι πολύ σημαντικό σε αυτήν εδώ την Επιτροπή θα είναι η συζήτηση που θα γίνει, η οποία θα είναι εις βάθος, ε, εμπαριστατωμένη και λίγα σημαντική. Θα συνεργαστώ ασφαλώς και με τον σκιώδη εισηγητή και άλλους συναδέλφους όσο καλύτερα μπορώ και αναμένω με μεγάλη ικανοποίηση αυτή την πρόταση για, ε, ως, ε, ως αυτή τη διαβούλευση, αυτή τη συνεργασία ως έναυσμα για την περαιτέρω πρόθεση του έργου. και ορισμένα μέλη της Επιτροπής είναι επιφυλακτικοί και δεν θέλουν ε, ένα μόνο άτομο να έχει συγκεντρωμένη στα χέρια του τόση πολύ εξουσία. Είμαι νέο μέλος και μέλος της νέας ομάδος της ECR και θέλω να συμβάλλω επικοδομητικά ως εισηγητής ξεπερνώντας τις κομματικές, τα κομματικά πλαίσια και θα μελετήσω με πολύ προσοχή ε, τις δυνατότητες χρηματοδότησης, πιστοποίησης γιατί θέλω Θέλω ο Γαλιλαίος να γίνει ένα πάρα πολύ επιτυχημένο πρόγραμμα ε, γι' αυτό προσβλέπω με ιδιαίτερη ικανοποίηση στη συνεργασία μαζί σας. Και γι' αυτό ε, με ικανοποιεί ιδιαίτερα η περαιτέρω συνεργασία μαζί σας. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρώτη σε αυτή τοποθέτηση. Η κυρία Τσικάου έχει ζητήσει το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την παρουσίασή του και να κάνω μια ερώτηση, αν μου επιτρέπετε, στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή της αρμόδιας αρχής. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας έχει στείλει ένα έγγραφο που δείχνει σαφή διαχωρισμό ανάμεσα στις διαδικασίες πιστοποίησης, μιλώ για θέματα ασφάλειας, δηλαδή ε, ένα συμβούλιο πιστοποίησης για την ασφάλεια από τη μια και από την άλλη έχουμε τις ε, δραστηριότητες ε, ε, σύμφωνα με το 683 του 2008. Αυτό τι προβλέπει. Ότι η διαχείριση και η διοίκηση όλων των θεμάτων ασφαλείας παραμένει στα χέρια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έτσι δεν είναι. Από την άλλη, ο πρόεδρος αυτού του Συμβουλίου εκπροσωπεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην αρμόδια αρχή θα μπορούσατε να μου απαντήσετε, να μου το ξεκαθαρίσετε αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Προς το παρόν δεν έχει ζητήσει το λόγο κανένας άλλος συνάδελφος. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να... Α, να απαντήσει η Επιτροπή μια στιγμή σε αυτή την ερώτηση και μετά θα συνεχίσουμε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ναι. Υπάρχει μια Επιτροπή Ασφαλείας που θέλουμε να συσταθεί, αλλά βασικά είναι μια επιτροπή των κρατών μελών αυτή. Είναι υψηλή αξιωματούχη ε, ασφαλείας των κρατών μελών. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με τη δική μας πρόταση, είναι ε, μέλος χωρίς δικαίωμα ψήφου στην Επιτροπή αυτή. Προφανώς οι αποφάσεις για την πιστοποίηση ασφαλείας είναι πάρα πολύ σημαντικές σε ένα πρόγραμμα σαν το Γαλιλαίο. Παράδειγμα, η Επιτροπή αυτή θα πρέπει να μας δίνει διέγκριση και άδεια για εκτόξευση, για ε, διαχείριση, για λειτουργία. Αυτά τα κάνουν ε, κατόπιν ε, επαληθεύσεις ότι έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα σύμφωνα με τις προαπαιτήσεις και τις προδιαγραφές ασφαλείας, την παραγωγή του εξοπλισμού. Όλα αυτά λοιπόν που είναι θέματα ασφαλείας. Πού θα γίνει το κέντρο εκτόξευσης, η πλατφόρμα, αν είναι επαρκής οι προδιαγραφές ασφαλείας, επαναλαμβάνω. Και από εκεί και πέρα δίνεται η έγκριση. Προφανώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρειάζεται εκεί για να δίνει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες στην Επιτροπή αυτή, πληροφορίες που χρειάζεται για να πάρει αυτές τις αποφάσεις. Και επίσης προτίθεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επισημαίνει ή να θέτει υπόψη αυτής της Επιτροπής κάποια σημεία που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ας πούμε, ε, αν είναι ένα θέμα ιδιαίτερα ακριβό ή αν προκαλέσει μεγάλες καθυστερήσεις. Είναι σημαντικό να το λέμε εμείς αυτό σε αυτή την Επιτροπή. Στο Συμβούλιο. Για να βλέπουμε από εκεί και πέρα πώς θα προχωρούμε. Και είμαι βέβαιος ότι και στην Επιτροπή σας εδώ θα γίνουν αντίστοιχες συζητήσεις. Πώς αλληλεπιδρούν τώρα όλοι οι πρωταγωνιστές του τους. είναι πολύ σημαντικό και αυτό. Χρειάζεται πολύ στενή συνεργασία και ε, ξεκάθαρη κατανομή και επιμερισμό αρμοδιοτήτων. Να ξέρει ο καθένα τι κάνει, γιατί είναι και πολύ σφιχτό το χρονοδιάγραμμα και πρέπει να προχωρήσουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Χολ, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Από το τελευταίο σχόλιο της Κομισιόν, την αλληλεπίδραση όλων είναι ιδιαίτερα σημαντικό, διότι το χρονοδιάγραμμα μας πιέζει. Μήπως θα μπορούσε η Κομισιόν να σχολιάσει το ότι ορισμένες χώρες μέλη δεν βλέπουν το πρόγραμμα αυτό με τον ίδιο τρόπο που τα βλέπει η Κομισιόν και το Κοινοβούλιο. Δηλαδή, ορισμένα κράτη-μέλη δεν θέλουν να έχει ρόλο παρατηρητή το Κοινοβούλιο στη νέα υπηρεσία. Επίσης φαίνεται να υπάρχει αντίθεση στο ρόλο της Κομισιόν. Να είναι δηλαδή πιο μεγάλος από ότι είναι το 50% του δικαιώματος ψήφου. Η Κομισιόν προβλέπει δυσκολίες στο σημείο αυτό. Μερικές κυβερνήσεις το θεωρούν ακόμα διακυβερνητικό πρόγραμμα όπως η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος ενώ εγώ έχω την εντύπωση ότι η Κομισιόν το θεωρεί περισσότερο κοινοτικό πρόγραμμα. Θα μπορούσε η Κομισιόν να μας πει ποια είναι η γνώμη της, τι πρέπει να γίνει από εδώ και μπρος έτσι ώστε ε, αυτές οι διαφορετικές απόψεις να εμποδίσουν την σωστή και έγκυρη εφαρμογή του προγράμματος. Ο κύριος Οντί Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ακριβώς το ίδιο μήκο κύματο με τη συνάδελφο Χολ. Αυτή η ιστορία με τον Γαγγιλέο είναι σαφής. Έχουμε δώσει 2 με 3 δισεκατομμύρια, δεν ξέρουμε όμως σε ποιον ανήκει ο Γαγγελέο. Έχουμε ένα κονσόρτιουμ ιδιωτικών επιχειρήσεων, μετά έχουμε μια αρχή, τώρα μας προτείνουν μια αζόνς, μια υπηρεσία φορέας. Ήμουν εισηγητής για το θέμα αυτό. Δεν είναι καν στους λογαριασμούς του 2007 της Ένωσης ο Γαλιλαίο. Πρέπει να τα ξεκαθαρίσουμε αυτό, να ξέρουμε τι θα είναι λειτουργικά ο Γαλιλαίος. Όσον αφορά το Διοικητικό Συμβούλιο, αν δούμε τα έγγραφα, από ό,τι φαίνεται, έχουμε μία διακυβερνητική δομή εδώ. Αν η Κομισιόν, όπως έκανε και στο παρελθόν, εξακολουθήσει να συμπεριφέρεται ως Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου, έχοντας το 50% των ψήφων και τα κράτη-μέλη το 50% και εμείς παρατηρητές. Εμείς δηλαδή ευρωβουλευτές ουσιαστικά δίνουμε μια εγγύηση κατά κάποιο τρόπο στο κοινωτικό αυτό πρόγραμμα χωρίς να έχουμε συγκεκριμένο εκτελεστικό ρόλο στο Διοικητικό Συμβούλιο. Και προσθέτω, υπάρχει ένα άλλο ερωτηματικό μεγάλο με όλε αυτέ τι υπηρεσίε που δημιουργούμε. Ένα σωρό υπηρεσίε δημιουργήσε η Ένωση. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό εδώ, αυτή εδώ η υπηρεσία. Ε, λοιπόν, πρέπει η Κομισιόν να διασφαλίσει το Κοινοβούλιο ότι θα έχουμε δικαίωμα πολιτικής παρακολούθησης της λειτουργίας αυτή της υπηρεσίας. Και επειδή είμαι και στην Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου, ελέγχου του προπολογισμού μάλλον, που θεωρείται ουδέτερη επιτροπή, προσθέτω ότι υπάρχει μία παράγραφο για τον έλεγχο του προπολογισμού όσον αφορά τη λειτουργία αυτή τη Υπηρεσία, διότι έχουμε μεγάλα προβλήματα στο να ελέγχουμε ένα σωρό υπηρεσίες. Πρέπει λοιπόν το σημείο αυτό να ξεκαθαριστεί στη συζήτησή μας. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ρενό. Ζωκίνα, ευχαριστώ πρόεδρε. Αν μη τι άλλο, μετά από όλα αυτά που ακούσαμε από τους δύο προλαλήσαντες, χρειαζόμαστε διευκρινήσεις. Το πρόγραμμα αυτό καθυστέρησε πολύ και κατά την άποψή μας είναι απολύτως απαραίτητο για τη στρατιωτική, οικονομική και πολιτική ανεξαρτησία της Ευρώπης από τις Ηνωμένες οι καθυστερήσεις, οι ολιγορίες και τα σφάλματα ε, οφείλονται σε πολιτική βούληση. Ορισμένα θέλουν να παραμείνουν ε, υπό το ζυγό των ΗΠΑ για λόγους ιδεολογικούς, για λόγους οικονομικούς, έτσι ώστε οι ιδιώτες και φιλελεύθεροι να διαχειρίζονται το πρόγραμμα. Είμαστε υποχρεωμένοι να διαπιστώσουμε ότι ε, σε όλα τα προγράμματα δημόσιου συμφέροντος που χρειάζεται χρόνο και ο Γαλιλαίος απέδειξε ότι δεν μπορεί να είναι ε, η διαχείρισή του ιδιωτική. Για να σώσει λοιπόν το φάκελο η Κομισιόν αποφάσισε να κοινωνικοποιήσει τις απώλειες, τις ζημίες. Αυτό δεν είναι πρωτοφανές αλλά ε, ε, είναι ας πούμε κάτι καλύτερο από την πλήρη εγκατάλειψη όπως θα ήθελε το αμερικανικό λόμπι. Εμείς δεν θέλουμε τώρα, εφόσον έχουμε ε, κοινωνικοποιήσει τις ζημίες, να ιδιωτικοποιήσουμε τα κέρδη του Γαλιλαίου. Χρειάζεται έλεγχος, έτσι ώστε η κοινωτικη προτίμηση να λειτουργεί και να ε, εκτοξευθούν οι δορυφόροι από την Αριάν και οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις κατά πρώτο λόγο να υποφεληθούν από τις επενδύσεις του Γαλιλαίου. Έτσι, με αυτόν τον προσανατολισμό θα έχουμε υψηλή ε, κοινωνική ποιότητα θέσει απασχόληση στην Ένωση και θα πρέπει να είναι και ένα σημαντικό εργαλείο χειραφέτηση τη Ένωση από το ΝΑΤΟ και τι Ηνωμένε Πολιτείε. Ευχαριστώ θερμά. Ο Σόζα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να σας πω μόνο ότι άκουσα με μεγάλη προσοχή ε, τα όσα μας παρουσίασαν σχετικά με αυτό το νέο πρόγραμμα και χαίρομαι που τα άκουσα αυτά γιατί είναι και σημαντικά και αξιοσημείωτα. Θα ήθελα όμως να σας εκφράσω μια ανησυχία που έχω γιατί είναι υπερβολικά βαριά η γραφειοκρατική δομή και οργάνωση και πολύ περίπλοκη κάθε προσπάθεια που καταβάλλεται για να διευκολυνθεί η κατάσταση και να είναι πιο απλή η διαχείριση αυτών των προγραμμάτων είναι πάντα ευπρόσδεκτη. Γιατί μία από τις κριτικές που ακούμε διαρκώς από τους Ευρωπαίους πολίτες είναι ακριβώς αυτό. Δηλαδή, ότι είναι τεράστια η περιπλοκότητα, ε, πυκνότητα και η γραφειοκρατική και η οργανωτική στους ε, ευρωπαϊκούς θεσμούς και τα θεσμικά όργανα. Εγώ λοιπόν είμαι υπέρ όλου αυτού του προγράμματος, αλλά με την προϋπόθεση ότι από οργανωτικής πλευράς θα είναι απλό και εύκολο. Και υποστηρίζω και αυτό που ακούσαμε προηγουμένως για τη συμμετοχή του Κοινοβουλίου στη διακυβέρνηση αυτού του προγράμματος και το Κοινοβούλιο πρέπει να παίζει ένα ρόλο πολύ πιο πρωταγωνιστικό από αυτό που του επιφυλάσσει το έργο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελε η Κομισιόν να απαντήσει και να συμπληρώσει. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τα μέλη για τις παρατηρήσεις που έκαναν. Θα πω λίγα λόγια μόνο. στις συζητήσεις που γίνονται τώρα στο Συμβούλιο είναι αλήθεια ότι τα κράτη, τα κράτη-μέλη δεν συμφωνούν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να έχει ένα μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο της, ε, του οργανισμού. Εγώ δεν μπορώ να πω την προσωπική μου γνώμη, θα αποφασίσουν τα θεσμικά όργανα. Αλλά ο ρόλος της Κομισιόν αυτή τη στιγμή ε, με το Συμβούλιο για το αν θα έχει μία θέση στο Συμβούλιο, στο Διοικητικό Συμβούλιο ή όχι. Εμείς είπαμε ότι είμαστε υπεύθυνοι για τα προγράμματα και εφόσον αυτό ισχύει τότε θα πρέπει να έχουμε και μία ουσιαστική επιρροή στη, στο Διοικητικό Συμβούλιο του TSA για να υπάρχει συνέπεια σε όλο αυτό το πρόγραμμα και στο χρονοδιάγραμμα και στο περιεχόμενο. Εάν δεν έχουμε μια τέτοια επιρροή, τότε δεν θα μπορέσουμε να παραδώσουμε το έργο αυτό εγκαίρως και μέσα στα πλαίσια του προϋπολογισμού ε, και δεν θα μπορέσουμε να είμαστε υπεύθυνοι για τις εργασίες της υπηρεσίας αυτής ξέρω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα ήθελε να έχει μία, να ακουστεί η φωνή του δηλαδή στην ανάπτυξη αυτού του προγράμματος, αλλά δεν νομίζω ότι είναι έτοιμο ακόμα. Εάν κάποιο όργανο είναι έτοιμο, αυτό είναι η Κομισιόν, η Εκτελεστική Επιτροπή. Γι' αυτό θα πρέπει να διευκρινίσουμε τι σημαίνει ουσιαστική επιρροή ε, για να μπορέσουμε να αποφασίσουμε ε, ποιος θα έχει εκπροσώπηση στο Διοικητικό Συμβούλιο. Αυτό θα το συζητήσουμε βεβαίως με εσάς και με τα άλλα θεσμικά όργανα. Διαφωνώ με ορισμένα σχόλια που ακούστηκαν όσον αφορά την περιπλοκότητα της δομής. Εγώ νομίζω ότι η δομή όλου αυτού του έργου είναι αρκετά απλή. Υπάρχει το όργανο, η βασική δομή για τη λήψη των αποφάσεων, το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε διαβούλευση με την Κομισιόν. Εν συνεχεία, η ευθύνη για την εκτέλεση είναι αποκλειστικά στα χέρια της Κομισιόν ε, ε, εκτός από μία πτυχή, ένας τομέα που είναι η πιστοποίηση. Η διαδικασία πιστοποίησης γίνεται πάντοτε ξεχωριστά από την εκτέλεση του προγράμματος προγράμματος έτσι ήθιστε και γι' αυτό δεν έχουμε ε, κανένα πρόβλημα ε, με τις εργασίες, με το έργο του, του GSE. Είναι δικές του, δικές του θα είναι οι υπηρεσίες ασφάλειας και θα είναι υπεύθυνο για τα προγράμματα τα οποία εκτελούνται στο, στο δικό του τομέα. Πιστεύουμε λοιπόν ότι η διάρθρωση είναι πάρα πολύ καλή έτσι όπως έχει συνταχθεί. Χρειάζομαστε μια ξεχωριστή υπηρεσία πιστοποίησης. Εκτός τούτου θα λειτουργεί το κέντρο ασφαλείας το οποίο θα είναι πάρα πολύ σημαντικό για να είναι ένα κέντρο σύνδεσμος με τα κράτη-μέλη για να συζητάει με, όλα τα, με όλους ενδιαφερόμενους τα θέματα ασφαλείας στο μέλλον και είμαστε βέβαιοι ότι αυτή η διασύνδεση με τα κράτη-μέλη είναι λίγα σημαντική αλλά και από πλευρά τη ευρωπαϊκή κοινότητα θα πρέπει να εξασφαλίσουμε το GSA θα έχει το κατάλληλο προσωπικό και τα κατάλληλα κονδύλια για να λειτουργήσει. Δεν, και επίσης δεν είναι δυνατόν να λειτουργήσει αν η ασφάλεια του συστήματος δεν βρίσκεται υπό πλήρη έλεγχο μία άλλη ερώτηση αφορούσε κύριο, ε, την, την, ε, και που ανήκει αυτό νομίζω είναι σαφέστατο τα προγράμματα ανήκουν στην κοινότητα τα, τα ενεργητικά ε, ενσωματώνονται, ανήκουν στον προϋπολογισμό της κοινότητας και εκτός από από ορισμένα κτίρια τα οποία έχουμε και ορισμένα τμήματα της υποδομής όλο το budget εμπίπτει στην κοινότητα. Είναι καινούριο στοιχείο και μεγάλο στοιχείο. Γι' αυτό πρέπει να γίνει σωστά η διαχείριση, η καταχώρηση και είναι σαφές ότι τα προγράμματα αυτά δορυφορικής ραδιοπλοήγησης ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την κοινότητα που φέρει και την ευθύνη του συστήματος. Νομίζω, Πρόεδρε, ότι απάντησα στις ερωτήσεις και... Είμαι ε, στη διάθεσή σας για να συζητήσω με την Επιτροπή σας ε, το θέμα αυτό στο μέλλον. Θα ήθελα να δώσω εν κατακλείδη το λόγο στον εισηγητή. Ευχαριστώ. Ακούσαμε πολλά σχόλια και θα πρέπει να επανέλθουμε ε, στις μελλοντικές μας συζητήσεις σε αυτό το θέμα. Δεν έχω τίποτα να προσθέσω τώρα. Πιστεύω ότι πολλά ελέγχθησαν και όλα αυτά θα ληφθούν υπόψη στην σύνταξη της εξέσεως. Ευχαριστώ και την Κομισιόν για την ε, προσέγγιση της και για την θετική στάση για την επίλυση των προβλημάτων. Ευχαριστώ πάρα πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Ολοκληρώσαμε το σημείο 4 το οποίο βεβαίως ε, θα συνεχιστεί η συζήτησή του, έχω την εντύπωση ότι το θέμα του Γαλιλαίου είναι τόσο σημαντικό και πολλοί συνάδελφοι έχουν κάνει ορισμένες παρατηρήσεις. Θα πρέπει λοιπόν να σκεφτούμε εάν μπορέσουμε στο μέλλον να κάνουμε μια ουσιαστική συζήτηση και για το Γαλιλαίο με την ευκαιρία αυτής εδώ της γενικής συζήτησης Συζήτηση του 4. Ε, καλό θα ήταν να κάνουμε αυτή τη συζήτηση τώρα που δεν έχουμε ακόμα έναν όγκο κειμένο, ε, μια μεγάλη τεκμηρίωση ε, στα γραφεία μας. Γι' αυτό θα ήθελα το, τη γραμματεία να εξετάσει αυτό το θέμα. Πότε πρέπει να κάνουμε μια συζήτηση σε βάθος για τον Γαλιλαίο. Ωραία, ολοκληρώσαμε λοιπόν την ημερήσια διάταξη σήμερα, το οποίο είναι ένα θαυμάσιο γεγονός. Σας ευχαριστώ για την πολύ πειθαρχημένη συζήτηση και εάν, εάν τα καταφέρουμε. Σας θέλαμε να καλέσουμε τους συντονιστές τώρα για να ε, προτάξουμε τη συνεδρίαση αυτή. Ελπίζω να μην έχει κανείς αντίρρηση. Εγώ δεν έχω. Πέντε λεπτά διάλειμμα να μήπως βρούμε τους συντονιστές.